Colleghi, per favore, prendete posto. I relatori sono presenti. Diamo inizio. Καθίστε, παρακαλώ, είναι εδώ οι συγητές. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε... 12 και 13 είναι οι συνέπειες τη ένταξης, της θέσης εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεν ξέρω πώς οργανωθήκατε κυρία Γκάλ, κυρία Λόχμπιχλερ. Ποιος θα μιλήσει πρώτος, η κυρία Λόχμπιχλερ. Είστε πρώτοι, σας ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην τελευταία μας συνεδρίαση της ΑΦΕΤ στις αρχές του Νοεμβρίου υποβάλαμε το σχέδιο έκθεσής μας. Οι τροπολογίες μας αφορούσαν διαφορετική διαδικασία επιτροπολογία για την υιοθέτηση του εγγράφου στρατηγικής με βάση το EIDHR. Αυτή η διαδικασία εξέτασης θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για μέτρα που εκπίπτουν των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που κατοχυρώνονται από την νομική βάση. Είχαμε εμβριθεί συζητήσεις για το θέμα αυτό και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια συνέπεια και συνάφεια από την πλευρά του Κοινοβουλίου η διαδικασία του RPS θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Κάτι που δίνει και βάση αλλά και συνέπεια και συνοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιχειρηματολογήσει σε μελλοντικέ διαπραγματεύσεις για μηχανισμούς εξωτερικών σχέσεων. Κάτι που είναι σημαντικό, μια και το ισχύον μηχανισμός θα εκπνεύσει το 2013. Επίσης, ε, θέλουμε πριν τις... ζητήσαμε πριν τις 4 Δεκεμβρίου να ψηφίσουμε πριν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεδομένου όμως ότι αυτή η απόφαση δεν θα είχε νόημα πια, θα ήταν παροχημένη μετά την 1η Δεκεμβρίου, αποφασίσαμε τελικά να μην ψηφίσουμε. Τώρα, δυνάμει τη συνθήκη τη Λισαβόνα, το RPS δεν εφαρμόζεται πια. Αλλάζει το σύστημα για την εφαρμογή τη ε, ε, νομοθεσία προβαίνοντα σε διάκριση μεταξύ των ε, διαδικασιών εκχώρησης και των διαδικασιών ε, ελέγχου που αντικαθιστά την παρούσα διαδικασία ελέγχου. Αυτή τη στιγμή τα θεσμικά όργανα έχουν διαπραγματεύσεις για το να μεταφέρουν τη νέα διαδικασία σε νομοθετικές διατάξεις. Και μάλιστα η Επίτροπος Φεραίρο Βάλτνερ έλαβε επιστολή από τον κύριο Αλμπερτίνη για μέτρα κατά του ΚΔΕ σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση των στρατηγικών γράφων. Και μάλιστα έχουμε και μια εκτενή ανακοίνωση με νομικά επιχειρήματα που αντιβαίνουν στη βασική θέση της Επιτροπής. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το πώς θα πρέπει η νέα διαδικασία να μεταφερθεί σε νομικά κείμενα. Και δεν είναι ακόμη δυνατό να υποβάλουμε τροπολογίες ε, με βάση τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πρόκειται για εξαιρετικές ε, συνθήκες και περιστάσεις στη μεταβατική περίοδο μεταξύ των δύο συνθήκων και αυτό προτείνουμε σήμερα να μην ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Θα ήθελα όμω να ζητήσουμε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να μα αναθέσει εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων επί των αρχών του εγγράφου στρατηγική που θα πρέπει να θεωρηθεί ω ε, ε, νομοθετική πράξη μετά από εκχώρηση. Ε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει άλλωστε μεταξύ των θεσμικών οργάνων για τι νομοθετικέ διατάξει σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εν τω μεταξύ και πέραν τη συζήτηση των νομικών θεμάτων είχαμε άτυπη και πολύ γόνιμη συνάντηση με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά το έγγραφο στρατηγικής για το EIDHR και προσβλέπουμε στη σύσταση ενός επίσημου, μιας επίσημης ομάδας εργασίας για το ADHR υπό την αιγίδα της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συμφωνούμε επίσης να, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει πιο επίσημη άποψη μετά την ε, επίσημη επίδοση του εγγράφου στρατηγικής από το Μητρό Επιτροπολογίας και μετά να αποφασίσει για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λοπτήλερ. Ο κύριος Γκάλ θέλει να παρέμβει και να συμπληρώσει η κυρία Η Μπάρμπαρα είπε όλα τα σημαντικά για αυτό το περίπλοκο, την περίπλοκη νομική διαδικασία στην οποία είμαστε βουτυγμένοι. Θα ήθελα να εξηγήσω στους συναδέλφους ότι σε αυτή την έκθεση έχουμε δύο ομάδες τροπολογιών. Η πρώτη ομάδα αφορά την πρόταση της Κομισιόν και την υποστηρίζει την πρόταση αυτή της Κομισιόν. Να επιτρέψει όλες οι δαπάνες να χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό του μέσου αυτού. Ε, χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία της Κομισιόν και την υποστηρίζουμε. Η άλλη ομάδα τώρα τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στην, με την έκθεσή μας καθώς και από τους συναδέλφους της Επιτροπής Ανάπτυξης, έχουν σαν σκοπό να δώσουν περισσότερες εξουσίες στο Κοινοβούλιο και να μπορούμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, ό,τι γίνεται ε, στο έγγραφο στρατηγικής και στο ετήσιο ε, πρόγραμμα. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την, συζητάμε αυτό το, το θέμα της νομικής ανασφάλειας, γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη διατύπωση για το πώς αυτή η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο θα ονομάζεται στο μέλλον και πώς θα περιγράφεται με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, αφού τεθεί σε ισχύ. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχουμε την κατάλληλη διατύπωση, να το συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας και εν συνεχεία θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ε, για το στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ ε, συζητάνε περισσότερο τον μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας και εμείς συζητάμε αυτό το μέσο. Η Κομισιόν ετοιμάζει ένα έγγραφο στρατηγικής, το οποίο θα μας το υποβάλει επίσημα. Γι' αυτό λοιπόν, περιμένοντας αυτό το έγγραφο, ζητάμε να αναβληθεί η ψηφοφορία και ζητάμε την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Ξεκάθαρη η παρέμβασή σας. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Μπράτλερ, όχι, ο κύριος Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, σε ποιον θα το δώσουμε αυτό. Η εντολή αυτή θα πρέπει να δοθεί στους εισηγητές, στους εισηγητές. Νομίζω ότι αυτό ζητάνε οι εισηγητές. Ας σας ακούσουμε όμως. Έχετε δίκιο. Ε, η κυρία Κίνγκα Γκάλερ και εγώ ε, ζητούμε αυτή την εντολή. Um, uh, το μέσο σταθερότητας ε, είναι το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη, αλλά θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε ήδη. Αυτό το οποίο εξήγησε ε, ήδη κυρία Λόχμπίλερ για τις ομορφικές πράξεις μετά από εκχώρηση, κατά την άποψή μου καλύτερο θα είναι να τα δούμε όλα αυτά τα μέσα της ΑΦΕΤ από κοινού και όχι χωριστά και το ίδιο να κάνουμε και με το DCI, το Μέσο Αναπτυξιακής ε, Συνεργασίας και να δούμε αυτό το σημείο με Συμβούλιο και Κομισιόν γιατί νομίζω ότι θα είμαστε ισχυρότεροι αν τα δούμε όλα μαζί από κοινού και παρακαλώ να μας δώσετε κοινή εντολή για όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, η λύση που προτάθηκε μεταξύ των υπηρεσιών και των εισηγητών είναι καλή και νομίζω μπορούμε να δώσουμε την εντολή αυτό το οποίο η συνάδελφος είναι πολύ χρήσιμο, δηλαδή να τα δούμε όλα αυτά μαζί και θέλω να ευχαριστήσω ε, όλους όσους εργάστηκαν για να βρουν μια λύση γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολο και προφανώς. Μούνιτσε e και Μπρόκ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω και ηγήτρια των Σοσιαλιστών, Πιστεύω ότι η προσέγγιση των δύο συγκεκριών για τα διάφορα μέσα σταθερότητας ε, είναι πολύ σωστή και θα εξασφαλίσει και το δικαίωμα ελέγχου μας. Με τους κανονισμούς αυτούς ουσιαστικά ανακτούμε αυτά που είχαμε χάσει στην πρώτη παρουσίαση των κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από χρόνια. Έχουμε πια ανακτήσει τον έλεγχο στα, στις ομοθετικές που μετά από εκχώρηση θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρί κανένα πρόβλημα λοιπόν, στενιζόμαστε την προσέγγιση των εισηγητριών. Ο κύριος Μπρόκ. Συμφωνώ με τους στόχους που αναφέρθηκαν και με τον στόχο της διαπραγμάτευσης εδώ πέρα της ε, κοινής. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνουν τα πράγματα αυτά στην αρχή αυτής της ε, περίοδου ισχύω των χρηματοδοτικών ε, μέσων αλλά ήταν ένα ευρύτατο σώμα εκεί όπου συζητήθηκαν όλα αυτά και τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να το συζητήσει μία μόνο κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να έχουν οι πράσινοι παντού τον, τον εισηγητή. Νομίζω πως η διαπραγματευτική ομάδα πρέπει να είναι λίγο πιο διευρυμένη για να εκπροσωπείται και αυτή η Επιτροπή. Ε, Μάλιστα. Λέζινγκ. Και μετά θα σας δώσω το λόγο, κυρία Λοχμπίλερ. Πρώτα, η κυρία Λέζινγκ. Ε, εσείς μίλησατε ήδη. Ας μίλησε και κάποιος άλλος πρώτα. Άσε. Ως ε, σκιώδης των ε, αριστερών, συμφωνώ με τα επιχειρήματα των ε, συναδέλφων. Χτες το συζητήσαμε αρκετά και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ότι αναλύσαμε τελικά αυτή την τόσο περίπλοκη κατάσταση. Μπίλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας στον κύριο Μπροκ, δεν είναι μόνο μία ομάδα που ασχολείται με αυτό. Ο κύριος Μίτσελ είναι στο άλλο μέσο, η κυρία Κίνγκαγκάλ είναι η συν ε, εκπρόσωπος και ο κύριος Σόιντς το αριστεράς είναι από την Ίντε και ο κύριο Μίτσελ είναι από την ΔΕΒΕ, την Επιτροπή Ανάπτυξης. Η κυρία Κίνγκεγκαλ ε, είναι και από την δική σας ομάδα. Αλλά εάν θέλετε να ενισχύσουμε την εικόνα του Κοινοβουλίου με ένα ακόμα άτομο, βεβαίως δεν θα έχουμε πρόβλημα και ακριβώς από τους ε, σοσιαλιστές θα μπορούσε να είναι. Εμείς είχαμε προγραμματίσει να διαπραγματευτούν οι συγητές με όλους τους ε, σκιώδεις, το είχα γράψει αυτό και χτες και έλεγα ρητός πως ε, καλό είναι να γίνουν οι διαπραγματευτικές προτάσεις και με εισηγητές και με σκιώδεις εισηγητές. Δεν ξέρω εάν θεωρεί ο κύριος Μπρόκ πως αρκούν οι οι εισηγητέ και οι σκιώδει εισηγητές ή να έχουμε περισσότερους. Εγώ νομίζω με εισηγητέ και σκιώδει τα, τα βολεύουμε. Αλλά δεν ξέρω τι άποψη έχει ο κύριος Μπρόκ. Πριν... Α, ναι, όχι, ο κύριος Μπρόκ τελικά. Και μετά Γκάλ και η Λυπή. Παρακαλώ. Εγώ πάντα έχω προβλήματα με τις σκιές και τους σκιώδεις, αλλά όχι σε αυτή την περίπτωση. Εάν είναι αυτή η λύση, θα το συζητήσουμε ακόμη μια φορά. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι σκιώδεις. Πρέπει να, να ρίξω μια ματιά. Αλλά εντάξει, αν είναι και οι σκιώδεις εκεί, ε, μπορούμε να το λύσουμε έτσι. Το legal, αλλά Αλλά το λόγο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τους σκιώδεις. Εγώ είμαι συνεισηγήτρια και και εγώ στην προηγούμενη συνεδρίαση είχα αρχίσει να παρουσιάζω την έκθεση. Τώρα συμφωνήσαμε με την κυρία Λόχμπίλερ ε, ότι εκείνη θα αρχίζει να παρουσιάζει το θέμα ως συνεισηγήτρια. Γι' αυτό άρχισε σήμερα η κυρία Λόχμπίλερ, αλλά είμαστε ισότιμες, ε, συντονιζόμαστε και συμφωνούμε σε όλα όσα είπαμε. Και ο κύριος Μίτσελ επίσης ε, παρακολουθεί στην άλλη επιτροπή αυτό το θέμα. Εγώ το παρακολουθώ εδώ σε αυτή την επιτροπή, την επιτροπή ΑΘΕΤ. Επομένω, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Ε, Ωραία τότε. Και μετά τα αυτά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι... Μισό λεπτό σας θυμάμαι. Ας ακούσουμε τους πάντες και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Μουνή. Eh, Ευχαριστώ. Το ΕΛΚΑ έχει δύο συντονιστές, εξού και τα προβλήματα. Δεν ξέρουν καν είναι οι συγγητές ε, των δύο εκθέσεων με εκπλήσει αυτή η κατάσταση να αναθέτουν σε δύο συντονιστέ αυτό το έργο του συντονισμού. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι η κυρία Μπράτνερ έλαβε υπόψη τη θέση των σοσιαλιστών σε ό,τι αφορά την κατάρτιση τη έκθεση. Γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το να διορίσουμε σκιώδη συγκητή, γιατί αυτό ήθισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, εντάξει. Μια και συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν έχουν ήδη μιλήσει. Ας ακούσουμε και τον κύριο Μίλλερ. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Όπως ανέφερε η κυρία Λοχ Μπίλερ, η Επίτροπος ε, Βάλτνερ σας έγραψε και σε εσά και στους συναδέλφους σας και είπε ποια, ποιες είναι οι θέσεις μας για τεχνικά θέματα. Ελπίζω αυτή η επιστολή να δοθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων η κυρία Βάντερ λέει στην επιστολή τη ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να διευκολύνει τι συζητήσει σα με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορούμε. Θα θέλαμε ε, να εκδοθεί γρήγορα ένα ψήφισμα για αυτό το θέμα Καλωσορίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία να δοθεί εντολή στους εισηγητές να συναντηθούμε το Συμβούλιο. Νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό τα δύο, οι δύο βραχίονες του νομοθετικού σώματος να αποφασίσουν για αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατόν και η Κομισιόν από την πλευρά της θα σας βοηθήσει όσο μπορεί στις συζητήσεις σας αυτές. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στα εξή ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξαχθούν από τις τρεις εισηγήτριε που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και μια εποπτεία από την Προεδρία αυτής της Επιτροπής. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει και ένα συντονισμός με τους κοιόδης ε, εισηγητές ε, μέσα σε ένα διευρυμένο πλαίσιο. Και αφού έχουμε καθορίσει ποιο είναι ο προσανατολισμό μα, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε εντολή για τι διαπραγματεύσει. Και να κάνουμε και τις, ε, στην τελική φάση τις απαραίτητες αλλαγές. Η κυρία Χάουτελα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή η λύση είναι καλή. Αλλά οι πολιτικές ομάδες δεν μπόρεσαν να, να ορίσουν τους συντονιστές τους που θα ασχοληθούν με το μέσο αυτό. Εγώ είμαι πρόεδρος ομάδας εργασίας που ασχολείται με το θέμα αυτό και με ανησυχεί το ότι δεν έχουν οριστεί ακόμη εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, γιατί θα προλάβουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Αν οι πολιτικέ ομάδε δεν ορίσουν του εκπροσώπου του για την εξέταση αυτού του θέματο, δεν θα προλάβουμε. Ελπίζω οι σοσιαλιστέ και το ΕΛΚ να φροντίσουν το συντομότερο δυνατό να ορίσουν του αρμοδίου, γιατί δεν μπορούμε συνέχεια να εργαζόμαστε άτυπα. Ναι, το ξέρουμε αυτό το επιχείρημα. Και αυτό που λείπει, γιατί Έχουμε καθορίσει τον προσανατολισμό και το πλαίσιο. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι τα ονόματα των ανθρώπων. Το καθήκον μου τώρα είναι να κινητοποιήσω τα, τις πολιτικές ομάδες, το Προεδρείο μαζί με τους συντονιστές, να προτείνουν λοιπόν κάποιους ανθρώπους. Κυρία Γκάλ. Κι εγώ υπάρχω. Υπάρχει το δικό μου όνομα στην όλη διαδικασία. Ήμουν από την αρχή εκεί όταν πρώτο ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΛΚ ε, μπορεί να με δώσει όνομα, αλλά εγώ ήμουν παρούσα, άρχισα τις διαπραγματεύσεις, δεν φταίει το ΕΛΚ. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι γίνεται εδώ πέρα. Πάντως, εμείς είμαστε εντάξει. Αρχίσαμε όπως έπρεπε και ήμουν παρούσα στην ε, εναρκτήρια συνεδρίαση όταν πρώτο ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει. Κανένα δεν επιρρύπτει ευθύνε, κυρία Γκάλ. Στην ομάδα στην οποία ανήκουμε. Νομίζω ότι είχα καταλήξει σε αποδεκτά συμπεράσματα. Είναι η τελευταία παρέμβαση, κυρία Μουνίθε. Εντάξει, είστε τελευταία που θα πάρει το λόγο οι σοσιαλιστές, οι σκιο... στους σοσιαλιστές, οι σκιώδεις συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ωραία. Τότε τελειώσαμε αυτό το σημείο στη μέση διάταξη. Το διεκπαιρεώσαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του ε, ενεργειακού ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο, ο κύριος Σάριους Βόλσκι μου ζήτησε να αναβάλουμε την ε, παρουσίαση της έκθεσής του, γιατί θα έρθει καθυστερημένα. Ο κύριος Λάσμπορφ κανονικά θα πρέπει να είναι εδώ, αλλά δεν τον βλέπω. Ο κύριος Λάμστορφ. Τότε ας περάσουμε στο τελευταίο σημείο στη μέση διάταξη. Την ετήσια έκθεση 2008 για την ΚΕΠΑ. Να σας δώσω κάποιες ενδείξεις για το πώς συντάχθηκε αυτή η έκθεση. Πρόκειται για μια ανταλλαγή προκαταρτικών απόψεων και η πιο ενδελεχή συζήτηση θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο. Το ψήφισμα καθορίζει κάποιες στρατηγικές, δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες, δεν είναι εξαντλητικά τα όσα αναφέρονται εδώ, συγκεντρώνεται στα πιο κύρια στοιχεία του θέματος. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης, με την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά μια νέα διάσταση, πολύ σημαντική. Επομένως, κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, μια συνεπή εξωτερική πολιτική. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει μια εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει απαραίτητους πόρους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο εγγυητής της ε, δημοκρατικής νομιμότητας εξωτερικής δράσης και θα πρέπει προφανώς να εμπλακεί άμεσα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΚΕΠΑ. Ο ύπατος εκπρόσωπος, που είναι η θεσμική καινοτομία της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, προσκαλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι κατ' εξαίρεση, αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε μια δομή. Επίσης, θα πρέπει να έχετε σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον διορισμό της διπλωματικής υπηρεσίας των ε, ειδικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία αναφέρονται τα αντικειμενικά διαφανή κριτήρια για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζεται εκ νέου ότι έχει μια μεγάλη ευθύνη σε ό,τι αφορά την ε, ευρωπαϊκή πολιτική κοινή ε, ασφάλειας. Στην έκθεση αυτό τονίζεται σε πολλά σημεία και τονίζεται ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τις διαθεσμικές ε, συμφωνίες που υπάρχουν σήμερα, ιδίως τη συμφωνία για την πρόσβαση στα εμπιστευτικά έγγραφα. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία επίσης σε μια διάσταση αποτελεσματικού σε μιας αποτελεσματικής πολυμέρειας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε επικοδομητική σχέση με τον ΟΗΕ και επομένως οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον ΟΗΕ, στη Γενέβη και την ε, Νέα Υόρκη θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα μέσα, πόρους, εργαλεία για να τα βγάλουν πέρα. Επίσης, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει μια δέσμευση απέναντι ε, στον διατλαντικό διάλογο. Επίσης, ε, στο ψήφισμα γίνεται μια ανάλυση των πολιτικών γραμμών σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θέματα όπως ε, ο Νότιος Κάφκασος, τα Δυτικά Βαλκάνια, το, το Αφγανιστάν και η Μέση Ανατολή. Επίσης, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο μεγάλο δυναμικό που έχει η εταιρική σχέση προς Ανατολάς και η Ένωση για τη Μεσόγειο. Στο παρελθόν το Συμβούλιο πάντα απέφυγε να παρέμβει στις ε, συζητήσεις της Επιτροπής για τις σχέσεις ε, και την ε, εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΚΕΠΑ. Με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας προσδοκούμε ότι είπα τος εκπρόσωπος που μας επιβεβαίωσε θα το κάνει, ελπίζουμε να το κάνει όμως κιόλα, θα εντοπίσει κάποιους διάβλους επικοινωνίας μαζί μας που θα συνιστούν πραγματικό διάλογο αυτό, έτσι συνοπτικά, είναι το περιεχόμενο της έκθεσης που σας προτείνω. Θεωρώ ότι όλοι σήμερα το πρωί ή χθε το βράδυ λάβατε το κείμενο μόνο στα αγγλικά. Τις επόμενες μέρες θα λάβετε και τις μεταφράσεις στις διάφορες γλώσσες. Και επομένως μπορείτε να παρέμβετε κι εσείς. Δεν ξέρω αν έχουμε ημερομηνίες για την υποβολή των τροπολογιών. Α, ναι. 12 Ιανουαρίου. 12 Ιανουαρίου. Μέχρι τις 12 υποβολή των τροπολογιών. Ανοίγει τώρα η συζήτηση. Eh, eh, allora, se Η σύντομη παρουσίαση που σας, έκανε, ε, που σας έκανα, σας άφησε άναυδους. Ε, ή μπορεί να λάβατε πολύ αργά το βράδυ χθε το κείμενο, Επομένω, μάλλον δεν προλάβατε να το διαβάσετε. Και άρα πώς να το σχολιάσετε. Α, υπάρχει κάποιος επιμελής, ο οποίος διάβασε το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και με συγχωρείτε που άργησα να σηκώσω το χέρι μου, δεν πρόσεχα στην τάξη. Όπως παλιά, στο σχολείο. Δεν έχω διαβάσει την έκθεση για να την κρίνω. Απλά να πω κάποιες ιδέες που νομίζω πρέπει να συμπεριληφθούν και νομίζω προέκυψαν μετά τη χθεσινή ακρόαση της Βαρόνης Άστον. Υπάρχουν ε, εδώ πέρα νομίζω διαφορές φιλοσοφίας μεταξύ κοινοτικής και διακυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να χαραχθούν κάποιες γραμμές ε, όσον αφορά την ε, λειτουργία της νέας αντιπρόεδρου της Κομισιόν και είπα της εκπροσώπου που βρίσκεται σε μια τελείως καινούρια κατάσταση. Οπότε πρέπει τώρα να παρέμβουμε, αλλιώς ε, θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Και εγώ ανησύχησα πάρα πολύ μετά τη χτεσινή ακρόαση, ας πούμε. Και αν είναι νομίζω να γράψουμε μια έκθεση μπορούμε να την κατευθύνουμε προς σωστή κατεύθυνση μέσω αυτής. Κύριε Μπρόκ, στη σύντομη εισαγωγή που έκανα, συνειδητοποίησα ότι δεν παρακολουθούσατε πολύ γιατί συζητήσατε την προηγούμενη έκθεση. Ε, κύριε Μπρόκ, όμως, αυτά που είπατε εγώ τα έχω αναφέρει ήδη. Θα τα δείτε πάντως και στην ίδια την έκθεση έτσι πιο αναλυτικά. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ούτε κι εγώ πρόλαβα να διαβάσω την έκθεση. Έφτασε και καθυστερημένα συνεδρίαση. Πιστεύω ότι η έκθεσή σας, θεματολογικά τουλάχιστον, αλλά και γεωγραφικά, καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα. Άλλωστε, πολύ σωστά η έκθεση επισημαίνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με βάση την ετήσια έκθεση. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και την ανάγκη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επί των αποφάσεων που αφορούν την ΚΕΠΑ, αλλά και την πολιτική άμυνας, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Το Συμβούλιο θα πρέπει να δείξει διαφάνεια για να δώσει και μια νομιμοποίηση στις ευρωπαϊκές πράξεις σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Καταρχήν, στην διατλαντική εταιρική σχέση και την έκκληση που απευθύνουμε προς την ύπατη εκπρόσωπο να προωθήσει μια σφαιρική προσέγγιση για τα διεθνή θέματα με τους Αμερικανούς εταίρους και μάλιστα χθες απέφθηνα σχετική έκκληση προς την κυρία Άστον και ζήτησα τη γνώμη της για το θέμα αυτό των διατλαντικών σχέσεων. Δεύτερον, κάνουμε μια θετική αξιολόγηση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κωσυφοπέδιο και τρίτον, υποστηρίζουμε την ανατολική εταιρική σχέση που είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Όντως, και αυτά τα επιχειρήματα καλύπτονται από την έκθεση. Ουσιαστικά υπογραμμίζεται επιχειρήματα που ήδη περιλαμβάνω στην έκθεσή μου και χαίρομαι που συμφωνούμε. Θέλει άλλος κανείς το λόγο? Ουδής. Οπότε ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και θα πρέπει προς στιγμή... Α, όχι, όχι, κυρία Μπραντνερ ζήτησε το λόγο. Συγγνώμη, δεν δε φαίνομαι εδώ πίσω. Ε, για την έκθεση συμφωνώ με τον κύριο Μπροκ. αυτά που ακούσαμε από την κυρία Άστον δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει με την εξωτερική υπηρεσία. Θα είναι στην Γενική Διεύθυνση Ρέλεξ ή θα πάει στα νέες αρμοδιότητες. Ε, το πού θα τοποθετηθεί αυτή η υπηρεσία στα νέε πολύ το συναρπαστικό. Δεύτερον, από πλευρά του Συμβουλίου υπάρχει ένα νέο έγγραφο για τις δυνατότητες ε, διαμεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το υποστηρίξουμε και να πούμε πως ε, θεωρούμε θετικό το ότι έχουμε νέες ε, κινήσεις σε έναν τομέα που είναι από τα ισχυρά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος στην, στις συμβάσεις με τρίτες χώρες, υπάρχει αυτή η γνωστή ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να αξιολογήσουμε το πώς λειτουργεί τελικά αυτή η ρήτρα κάπως πιο σοβαρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπράντνερ. Θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας και μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, όπως σας είπα, έχετε το χρόνο να καταθέσετε τροπολογίες που θα τις λάβω υπόψη. Δεν ζητάει άλλος κανείς το λόγο και προς στιγμή θα πρέπει να διακόψουμε γιατί οι δύο συγγητές μας, ο κύριος Άριος Βόλσκι και ο κύριος Λάμστορφ που είναι αρμόδιοι με τα, τις δύο επόμενες εκθέσεις ε, απουσιάζουν. Γι' αυτό ας κάνουμε μια δεκάλεπτη διακοπή περιμένοντας τους δύο εισηγητές μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ραντεβού σε 10 λεπτά.